Κυρία, κυρίες και κύριοι, Αλεσάνδρα Μορέτη παρετήθηκε, μου ανακοίνωσε δηλαδή ότι σταματά να είναι Ευρωβουλευτής από τις 2 Φεβρουαρίου του 2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραγράφους 1 και 3 του κανονισμού,